Λοιπόν, θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο Μπουλκ και την ε, Επιτροπή να μας ε, ανημερώσει για, ε, για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης ε, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στο Λονδίνο. Ε, θα μας μιλήσετε ειδικά για τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυσιπλοεία όσον αφορά την ε, εισφορά της, της ε, στη μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων της συνθήκης των Παρισίων. Θα ήταν χρήσιμο να δούμε πώς ε, μπορεί η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τις προσπάθειες της IMO προκειμένου να προβεί στην εκπλήρωση των στόχων αυτών. Και θα ήθελα επίσης να μας ε, μιλήσετε για την ε, ενημέρωση, ενημέρωση της ε, προσεχούς εφαρμογής της διεθνούς πολιτικής αλίας και την απαγόρευση των θαλασσίων αποβλήτων και των, της απόρριψης πετρελαίου στα, στη θάλασσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ε, βοηθήσατε για την επιτυχή διοργάνωση της ε, αποστολής μας στο Λονδίνο. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Πίτροπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Αντιπρόεδροι. και βεβαίως αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πράγματι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για δεύτερη φορά στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι εδώ για να σας ενημερώσω για την Συμφωνία Ορόσημο για, τους διεθνείς, για το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοεία, το Διεθνές Αριθμιστικό Όργανο. Όπως γνωρίζουμε, η διεθνής ε, ναυσιπλοεία αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των ε, στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση άσχε μεγάλη πίεση να ΑΕΜΟ για πολλά χρόνια και το θέμα αυτό κατάστηκε κατεπήγον όσον αφορά την αύξηση της θαλάσσιας ε, ρήπανσης. Η συνάντηση της ε, Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος ε, ενέκρινε την στρατηγική για την μείωση των ρήπων που αυξάνουν τα αέρια του θερμοκηπίου. Πρόκειται για την συμπερίληψη μιας, ε, του στόχου μείωσης των αερίων θερμοκηπίου κατά 50% το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 2008 με στόχο μακροπρόθεσμα την πλήρη ε, κατάργηση του άνθρακα ή δυνατόν αυτό τον αιώνα. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω σχόλιο εδώ, πιστεύω ότι τα επόμενα 30 χρόνια οι τεχνολογίες θα βελτιωθούν ε, σημαντικά, ούτως ώστε μπορούμε να αναμένουμε ε, ένα αποτέλεσμα μηδενικής ε, ρήπανσης ε, στον τομέα των μεταφορών. Αλλά να επανέλθω στην ΑΕΜΟ, είναι η πρώτη φορά που έχει συμφωνηθεί ένα στόχος μείωσης των ρίων του θερμοκηπίου για την αυσιπλοεία. Πιστεύω ότι και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, ελπίζω ότι μπορούμε λοιπόν να αναμένουμε φιλόδοξα προγράμματα ε, για την ε, ναυσιπλοή. This deal was not... Ελπίζουμε να ακολουθήσει και αεροπλοεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ήταν πραγματικά έπαιξε ένα ρόλο κλειδί προκειμένου να συμβεί αυτό. Όσο για σας που ήταν παρόντες εκεί ε, μπορούν να πιστοποιήσουν ότι πραγματικά αντιμετωπίσαμε μια σημαντική πρόκληση για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πολλές χώρες ε, αρχικά ήταν αρκετά πρόθυμες να συμφωνήσουν ε, για οποιαδήποτε ποσοτικοποίηση των εκπομπών και χάρη σε πολύ επιδέξιες διαπραγματεύσεις εκτός της αίθουσας συναντριάσεων και των ε, Προέδρων των Ομάδων Εργασίας και της Επιτροπής ε, επέφεραν ε, αυτό το αποτέλεσμα και έψαν την πλειονότητα των χωρών μελών του IMO. η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ έπαιξε σημαντικό ρόλο. Η Επιτροπή καθοδήγησε το συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ η, ίδια συνάντησα τις πράγματα αυτές από τις χώρες μέλη και τους έδωσα πλήρη υποστήριξη προκειμένου να μείνουν ισχυροί και ενωμένοι ε, εν ώψη αυτών των τόσο δυσχερών συζητήσεων. Και όλοι, και θα πρέπει να το τονίσω, όλοι ε, πραγματικά το έπραξαν. Ε, έδειξαν μεγάλο ζήλο και ήταν ε, οι 13 αυτές χώρες που διατύπωσαν την πλήρη τους υποστήριξη για την επίτευξη αυτών των στόχων. Και εγώ ως Επίτροπος ήμουν πολύ περήφανη που μπορέσαμε να συνενώσουμε τις προσπάθειές μας και να ε, οδηγηθούμε σε αυτά τα αποτελέσματα, σε αυτό το σημαντικό θέμα. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστώ και εσά τους ε, βουλευτές, τον κύριο Εκχάου, την κυρία Σουίτσα, οι οποίοι ήταν μέλη αυτή τη αντιπροσωπεία και έπαιξαν πολύ επικοδομητικό ρόλο οδηγώντα σε ε, ε, ε με τους εταίρους στην ΑΕΜΟ, συμπεριλαμβάνομενων και των επιχειρηματιών. Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερως περήφανη για αυτό το αποτέλεσμα, ε, το οποίο πέτυχε με, δημιουργώντας ένα συνασπισμό με τους τέρους μας στον κλάδο της ναυσιπλοποιίας ε, και τέλος ε, πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες όπως η δήλωση των Ιντεμπρούμ βοήθησαν να επιτευχθεί πολιτική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η αρχική στρατηγική του Α.Ε.Μ.Ο. είναι ένα ενθαρρυντικό πρώτο βήμα στον δρόμο αυτό τη ε, πλήρη ε, απομάκρυνση από τον άνθρακα. Αλλά υπάρχει μια γενική συμφωνία τη στρατηγική, η οποία υιοθετήθηκε στο Α.Ε.Μ.Ο. Είναι μια στέρεη βάση για μελλοντικέ ε, δράσει στον κλάδο αυτό. Η συμφωνημένη μείωση των εκπομπών αντιπροσωπεύει την αρχική εισφορά του Διεθνούς Κλάδου Αναυσπρολίας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των Παρισίων οι οποίοι μπορούν να αναθεωρηθούν στον το χρόνο. Και αυτό είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικό μια στιγμή, μια συγκυρία που βλέπουμε ότι οι υπολογισμοί που στο παρελθόν δεν ήταν πολύ ακριβείς και δυστυχώς πήγαιναν στη λάθος κατεύθυνση. Άρα λοιπόν μπορούμε ενδεχομένω η αύξηση της δημοκρασίας μας θέτει προ ακόμα σοβαρότερων απειλών. Ελπίζουμε λοιπόν όλοι να αυξήσουν τα επίπεδα των φιλοδοξιών τους ούτως ώστε να υπάρξει να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Είναι σημαντικό να υπάρξει καθοδήγηση προς τους βιομηχανικούς ε, κύκλους να αποστατικοποιηθούν οι στόχοι ε, προκειμένου να δοθεί ένα έναυσμα στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες με μηδενικά καύσιμα ε, από άνθρακα. Ελπίζουμε ότι η ανάπτυξη των σωστών τεχνολογιών ε, καθώς και η ανάπτυξη, εξέλιξη πράσινων ε, ε, πλοίων και καύσαμε με μηδενική ρήπανση, συνιστούν μια μεγάλη ελπίδα για το μέλλον και ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει αυτή την στρατηγική με πεπισμένη ότι καθώς ε, οδηγούμεθα στον δρόμο αυτό θα συνειδητοποιήσουμε τα ωφελήματα και καθώς και την εξοικονόμηση του κόστους. Η αρχική στρατηγική η οποία εγκρίθηκε παρέχει έναν ε, περιεκτικό κατάλογο βραχυπρόθεσμων, μέσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ε, μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Η στρατηγική επίσης επιβεβαιώνει ότι τα μέτρα τα οποία είναι εφαρμοστέα στα πλοία θα εφαρμοστούν με έναν τρόπο που να μην επιφέρει διακρίσεις ε, ε, και η στρατηγική εξασφαλίζει υποχρεωτικά μέτρα να είναι εφαρμοστέα στα πλοία και να εφαρμόζονται σε όλα τα σκάφη ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα από τη σημεία που φέρνουν. Επίσης, η στρατηγική αναγνωρίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της μείωσης των εκπομπών και ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ανάγκες των ετσόμενων χωρών, στα μικρά νησιά κλπ. Και στις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, χώρες. Η στρατηγική επίσης αναγνωρίζει υποστηρικτικά μέτρα για παράδειγμα μέτρα τεχνικής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της ε, ανάπτυξης, για την ανάπτυξη του δυναμικού και να γνωρίζει το ρόλο ε, του Διαχειριστικού Συμβουλίου της ΑΕΜΟ και των ε, κέντρων δικτύωσης και συνεργασίας που χρησιμοποιούνται ως προγράμματα αύξησης του δυναμικού μας και αρχίζουν να παράγουν τα πρώτα αποτελέσματα. Το επίπεδο των φιλοδοξιών ε, μπορεί βεβαίω να προωθηθεί περαιτέρω. Η στρατηγική επίση περιλαμβάνει ε, κάποιους ιστορικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν να αναθεωρηθούν παρά την αναθεωρημένη στρατηγική η οποία θα εγκριθεί το 2023 και αυτό μπορεί να γίνει εξετάζοντας τα δεδομένα για του υφιστάμενους ε, ρήπους ούτω ώστε να αναθεωρηθούν ε, σε σχέση με, τα, με που έχουν διατυπωθεί. Ε, θεωρώ ότι το πλαίσιο αυτό είναι καλό. Βεβαίως απομένουν πολλά πράγματα να γίνουν στο μέλλον και όπως άκουσα τα μηνύματα από το Κοινοβούλιο είναι θετικά και δεν μπορώ πάνω να συμφωνήσω. Ο θα πρέπει να συμφωνήσει επί ενός προγράμματος δράσεων παρακολούθησης προκειμένου να εφαρμοστεί η στρατηγική αυτή και χρειάζεται να υπάρξει μια συμφωνία ε, προκειμένου να προθεί η διαδικασία συμφωνίας για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Και αυτό είναι σημαντικό εάν θέλουμε ε, η ΑΕΜΟ να μπορέσει να υιοθετήσει αυτούς τους στόχους για το 2000, να πετύχει αυτούς τους στόχους το 2023. Ας αντιμετωπίσουμε λοιπόν το θέμα. Δεν πρόκειται τα πράγματα να είναι εύκολα. Έχουμε μείζονες προκλήσεις μπροστά μας. Υπολογίζω λοιπόν σε μια ε, στενή συνεργασία και ένα πνεύμα συνεργασίας προκειμένου ε, να έχουμε αποτελέσματα και μοντέλα πλήρους κλίμακας. Τώρα, ε, κατά κλείδι, θα ήθελα να σας ε, αναπτύξω κάποιες σκέψεις. Πιστεύω ότι με την έγκριση της ε, αρχικής στρατηγικής στο ΑΕΜΟ και ο Διεθνής Κλάδος Ναυσιπλοείας κατέδειξαν τη δήλωσή τους να αποτελέσουν κομμάτι της λύσης και νομίζω το μήνυμα αυτό είναι ήταν ξεκάθαρο και πραγματικά ήταν, ε, οφείλεται στις προσπάθειες του ΑΕΜΟ. Αλλά όπως είπα θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις προκειμένου να παράσχουν το πλαίσιο και τα συγκεκριμένα προγράμματα δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της ως ένας ισχυρός ε, παγκόσμιος ε, φορέας, ούτως ώστε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει να ελοπιθούν. Και δεν μπορώ παρά να σας διασφαλίσω ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί του σύναγκης την ε, πρόοδο προς την εκπλήρωση των στόχων μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και να θεσπίζει συνοδευτικά μέτρα ούτω ώστε ο τομέα να εισφέρει καθοριστικά στην επιτεύξη των στόχων των Παρισίων. Εάν ε, δεν έχει επιτεθεί ε, σημαντική πρόοδο το 2023, η Επιτροπή θα είναι η πρώτη η οποία θα προτείνει επαρκή δράση Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σήμερα Νομίζω ότι μπορούμε να δηλώσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Πετύχαμε μια καλή συμφωνία. Κατα... Προσπαθώντας να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλληλεγγύη. Και πριν κλείσω, επιτρέψατε μου εν συντομία να αναφερθώ σε τρία θέματα. Πρώτον, η έγκριση μέτρων που απαγορεύουν την μεταφορά ακατέργαστο πετρελαίου που δεν ε, συμφωνεί με το αποδεκτό όριο περιεκτικότητας σε θείο αναμένεται να ε, ληφθεί η σχετική απόφαση τον Οκτώβριο. Επίσης το ΑΕΜΟ συμφώνησε να συζητήσει την απαγόρευση για τη χρήση ε, το και την μεταφορά ακατέργαστου πετρελαίου στα, αρκτικά, στα ύδατα της Αρκτικής και τα δύο μέτρα είναι πολύ σημαντικά για την προστασία ενός πραγματικά αυθεντικού αρκτικού περιβάλλοντος που παίζει τόσο κρίσιμο ρόλο για το κλίμα μας. Τρίτον, θα ήθελα να τονίσω ότι το θέμα των θαλάσσιων αποβλήτων ε, λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερη προσοχή στον ΑΕΜΟ που ζήτησε υποβολή προτάσεων για να ε, την Μάρπολ ε, για να τα προωθήσει στη Μάρπολ και σε αυτό το πλαίσιο προσβλέπω στις επερχόμενες συζητήσεις για τη δική μας προτινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας που αφορά τις ειδικέ εγκαταστάσεις στα λιμάνια για την ρήψη των λιμάτων από τα πλοία έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των θαλασσίων λιμάτων και ε, αυτό στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Αυτά είχα να σας πω και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας απευθύνω το λόγο. Σας ευχαριστούμε και εμείς Επίτροπε για την ενημέρωση αυτή. Θα δώσω το, λόγο στα μέλη και πρώτα βέβαια θα ξεκινήσω με ένα μέλος που συμμετείχε στην αντιπροσωπεία και τους δύο συμπρόεδρους. Πρώτος λοιπόν ο κύριος Φαρία. Όχι. Η κυρία Γκούτελαντ πρώτα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Φαρία που μου δώσατε το λόγο. εγώ συμμετείχα σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της αποστολής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε, για την ε, μεγάλη σας προσήλωση. Ξέρω πως εργάζεστε σκληρά και εργαστήκατε σκληρά στη διάρκεια της διάσκεψης. Επίσης, ε, δείξατε την ε, αφοσίωσή σας στο θέμα και ενδιάμεσα. Και ευχαριστώ και ολόκληρη την ομάδα της Επιτροπής για τη σκληρή δουλειά που κάνει. Ξέρω πως ο συντονισμός των κρατών είναι πάρα πολύ σημαντικός στο Λονδίνο τα κράτη-μέλη έκαναν πολύ σημαντική δουλειά στη διάρκεια αυτής ε, της ε, συνόδου MEP ε, και επίσης πέτυχαν ένα μεγάλο βήμα πρόοδου. Ξέρουμε πως τα κράτη-μέλη θέλαν περισσότερα, ζήτησαν στόχο 70 με 100% μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 και ο τελικός στόχος είναι χαμηλότερος, ωστόσο εξακολουθεί να είναι μέγα βήμα μπροστά ε, ο καθορισμένος στόχος του 50% στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής και είναι και μια μεγάλη κίνηση το να υιοθετήσει μια στρατηγική ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το σημειώσουμε και να το επενέσουμε τον IMO για αυτό το βήμα μπροστά. Όμως ε, και είμαι ευτυχής που αναφέρατε πολύ ξεκάθαρο ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να ε, πιέζει, γιατί δεν αρκεί. Ήταν ε, λιγότερα αυτά που πετύχαμε από αυτά που χρειαζόμαστε αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε τις δεσμεύσεις του Παρίσιου. Επίσης, ο κόσμος της ναυτιλίας ξέρει πως ε, το πρόβλημα των εκπομπών από την αυτιλία, από την αυσιπλοεία ε, ε, διωγγώνεται και αν δεν μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική θα είναι μεγάλο το πρόβλημα όσον αφορά το διοξίδιο του άνθρακα. Το 2050 μπορεί να, η ναυτιλία να συμβάλλει κατά 70% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και μαζί με την αεροπλοεία είναι ο μεγαλύτερος ρηπαίνων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεχίσουμε να ασκούμε πίση και εσείς το περιγράψατε πάρα πολύ καλά διότι το 73 είναι σημαντική ε, χρονιά να ζητήσουμε σημαντικές δράσεις, σημαντικές ενέργειες πριν, αλλά θα υπάρξει και συζήτηση για το τι ακριβώς χρειάζεται, πόση δράση χρειάζεται. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2023. Πρέπει να ζητήσουμε στην επόμενη επίση να, να φέρει αποτελέσματα. Σας άκουσα που το είπα, η Κομισιόν πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη στο τι ζητάει, συγκεκριμένες δράσεις. Γιατί αν αφήσουμε να περνάνε τα χρόνια, δεν θα ε, καταφέρουμε να προλάβουμε αυτή την κατάσταση ε, που φοβόμαστε για το μέλλον, δηλαδή να είναι η ναυσιπλοή ένας από τους μεγαλύτερους ρηπαίνοντες στο μέλλον. Παρακαλώ λοιπόν την Κομισιόν συνεχίστε, μην σταματάτε την πίεση, ε, απειλήστε ε, για νομοθεσία και εμείς ως Κοινοβούλιο θα σας στηρίξουμε και θα συνεχίσουμε και από τη δική μας πλευρά τη σκληρή δουλειά. Γιατί αυτό το κάνουμε προς το συμφέρον της ε, πραγματοποίησης της συμφωνίας ε, του Παρισιού αλλά και για την ε, βιομηχανία της ναυσιπλοείας, το κλάδο μάλλον της ναυσιπλοείας γιατί αν δεν αλλάξει η τακτική θα μείνει μια πεπαλαιωμένη βιομηχανία πράγμα που δεν θα την βοηθήσει στο μέλλον. Στη διάρκεια της διάσκεψης λένε ε, άκουσα κάποιους να λένε ότι θα πρέπει οι υπόλοιποι να κάνουν την πρόοδο. Όχι, εκείνοι οι ίδιοι θα πρέπει να ε, φέρουν την τεχνολογική πρόοδο. Όπως πιέζουμε την αυτοκινητοβιομηχανία, όπως πιέζουμε την βιομηχανία, έτσι θα πρέπει να τους πιέσουμε και εκείνους. Δεν μπορούν να λένε ότι άλλοι θα κάνουν τη δουλειά στη θέση τους. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά εκείνοι θα πρέπει να παροτρύνουν το ίδιο του στον κλάδο και ε, να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την καλή μας συνεργασία. Ευχαριστώ κύριο Σφαρία. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Χαρά μας πάντοτε να σας βλέπουμε εδώ και ιδιαίτερα στις συνεδριάσεις με τον IMO που είσαστε ιδιαίτερα δραστήρια. Είστε πραγματικά ε, μια πολύ ισχυρή και προσιλωμένη προσωπικότητα που αγωνίζεται κατά των κλιματικών αλλαγών. Το ξέρουμε αυτό και είναι πάντοτε πολύ ε, θετικό να είμαστε μαζί σας. Ξέρουμε πως τονίζετε τη σημασία των φιλοδοξιών μας. Λέτε πως επετεύχθη καλή συμφωνία. Όπως και η συνάδελφός μας έλεγε, δεν είναι τόσο καλή το ξέρουμε μεταξύ μας. Και ε, είπατε ότι πρόκειται για συμφωνία ορόσημο στη διεθνή, στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και ότι ο ένας στόχος ποσοτικοποιημένος για την εκπομπή ε, αερίων του θερμοκηπίου που θα φτάσει στην μηδενική εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα το 2050. Όμως, ε, Πίτροπε, μην το λέτε αυτό γιατί δεν θα γίνει συγκρίναμε με το εκπομπέ του 2008 και τελικά κάτι τέτοιο δεν μπήκε στο τελικό κείμενο. Το απέφυγαν αυτό. Εμείς το θέλαμε αυτό. Όπως γνωρίζετε, Έχουμε τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Ναυσιπλοεία για το MRV και αυτό απαιτεί από τα πλοία που τα πλοία να ε, αναφέρουν τις εκπομπές τους. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει λοιπόν τη διαφάνεια στις εκπομπές και πραγματικά αποτελεσματικά στοιχεία για τους ευθύνοντες για τη συμπλήψη των πολιτικών αποφάσεων. Το ίδιο για την αυσιπλοή και για, το... για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ο ΑΕΜΟ έχει το δικό του σύστημα και λέγεται αυτό σύστημα συλλογής δεδομένων. Ένα νέο σύστημα, με αυτό το σύστημα μάλλον θα αναθεωρηθεί, αυτό ήδη έχει αναφερθεί και για να είναι ευθυγραμμισμένο με το σύστημα του IMO. Κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι πότε προγραμματίζει η Επιτροπή να φτιάξει την πρόταση για την αναθεώρηση ε, του κανονισμού και διασφαλίζεται η διαφάνεια στα πραγματικά στοιχεία περί φορτίων, περί ε, φορτηγών πλοίων. Γιατί αυτή είναι η πραγματικά, πραγματική διαφορά, ότι δηλαδή ε, τα πραγματικά στη δεδομένα για τα φορτηγά δεν υπάρχουν, γιατί διαφορετικά εμείς ευθυγραμμιζόμαστε μαζί τους προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Τέλος, η Κομισιόν θα υπερασπιστεί μια πιο προοδευτική, ξέρω ότι είστε πολύ προοδευτικοί σε αυτό το τομέα, πιο προοδευτικό, διαφανή και αποτελεσματικό κανονισμό ή θα το εγκαταλείψει υπέρ των χαμηλότερων φιλοδοξιών του IMO όσον αφορά τη συλλογή των δεδομένων θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ θετικό που ε, τουλάχιστον και επιτέλους ο ΑΕΜΟ κατέληξε κάπου στο θέμα που συζητήθηκε στην συνεδρίαση για την απαγόρευση των ακατέργαστου πετρελαίου στην Ανταρκτική. Για την Αρκτική όμως, για την Αρκτική δεν θα ισχύσει τέτοια απαγόρευση. Εγώ την περασμένη εβδομάδα συμμετείχα στο Παγκόσμιο Θαλάσσιο Πανεπιστήμιο και είχα τη χαρά να ρωτήσω τον εκπρός τους εκπροσώπους του IMO εκεί και δεν έλαβα απάντηση βεβαίως. Με αυτό τελειώνω και επανέρχομαι Ευχαριστώ όσο είπε η συνάδελφος, ότι η δικιά σα δουλειά είναι πολύτιμη και μας δίνει και εμά ένα κίνητρο για να είμαστε ακόμα πιο δραστηροί σε αυτά τα θέματα. Ξέρω πω είστε φιλόδοξοι και εμεί είμαστε φιλόδοξοι. Α πιέσουμε όσο γίνεται περισσότερο, χωρί βέβαια να σπάσουμε το σκηνή βέβαια, χωρίς να το παρατραβήξουμε. Να πω μόνο τέλο, Πρόεδρε και Επίτροπε, πω η συνάδελφο Σουίσα δεν μπορούσε να είναι παρούσα σήμερα, ήθελε, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Γι' αυτό και σας ζητά συγγνώμη που λείπει. Σας ευχαριστώ πολύ. Very πολύ. Ο κύριος Αϊκχάουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο. Καλώς ήρθατε. Πράγματι, και εγώ χάρηκα που σας είδα στο Λονδίνο και συμφωνώ με τους συναδέλφους που σας συνεχάρισαν και εσάς προσωπικά, αλλά και ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διαδραματίσατε τόσο σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας. Να προσθέσω εδώ και την Εσθονική Προεδρία που ασχολήθηκε με αυτό το φάκελο και ήταν χρήσιμο που ένα από τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ένιωθε ότι είχε την ευθύνη να προετοιμάσει το έδαφος ε, για την επιτεύξη της συμφωνίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και εν ώψη των επερχόμενων συνεδριάσεων, γιατί όσο πιο προετοιμασμένοι είμαστε, τόσο το καλύτερο θα είμαστε και πιο ενωμένοι, το οποίο δεν ισχύει πάντα, όπως ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν προκειμένου όμως πήγε πολύ καλά ε, και ως ε, μέρος ε, της, ε, του συνασπισμού αυτό θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Βέβαια και η Νίση Μάρσαλ έπαιξαν σημαντικό ρόλο εδώ και να το αναφέρουμε. Θα φτάσουμε στο τέλος στην αεροπλοεία. Δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη αυτό. Όμως φαίνεται ότι η πίεση σε έναν οργανισμό όπως ο IMO ε, αποφέρει καρπούς. Τελικά ένιωσαν αυτή την πίεση ότι πρέπει κάτι να παράξουν ως αποτέλεσμα. Γιατί κατάλαβα και εκείνη ότι δεν γίνεται να περάσει εβδομάδα χωρίς να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και νομίζω ότι αυτό ε, ε, ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο, γιατί μπορεί κανείς να έχει ένα συνασπισμό τέτοιο, αλλά τελικά στην πράξη να μην έχει αποτελέσματα. Όμως βλέπουμε ότι τελικά έχει εμπροκειμένο. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται. Κοιτάζοντα τα όσα κάναμε στο Λονδίνο, νομίζω ότι υπάρχει μια ανησυχία για τη Λατινική Αμερική. Πολλέ χώρες μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα μας παρουσιάσουν δυσκολίες. Σαουδική Αραβία, εντάξει, δεν προκάλεσε καμία έκπληξη ε, ή ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν ήταν πολύ αξιόπιστο εταίρο, ούτε αυτό ήταν έκπληξη, αλλά για τι χώρε τη Λατινική Αμερική. έχουν ορισμένε επιφυλάξει και προβληματισμού γιατί απέχουν περισσότερο από την παγκόσμια αγορά και το κατανοούμε. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στι σχέσει μα μαζί του για να κάνουν τα απαραίτητα βήματα. Κάτι τελευταίο. Είπατε ότι είναι συμφωνία ορόσημο. Από πλευρά IMO πράγματι είναι. Μετά από πλευρά ε, κλιματική, εντάξει, δεν είναι και τόσο ορόσημο. Από πλευρά IMO βέβαια ήταν πολύ χρήσιμος ο ρόλος ε, του κλάδου. Και ως πράσινοι εμείς πάντα ξέρετε ότι παραπονιόμαστε, αλλά κάποιες φορές είναι σημαντικό και να τους ε, συγχαίρουμε εκεί που τους αξίζει. Και αυτό σίγουρα ισχύει αυτή τη στιγμή έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας, γιατί είπαν ξεκάθαρα τις τελευταίες ημέρες ότι εμείς μπορούμε να δεχθούμε αυτή την ε, μείωση ε, των εκπομπών. Κάποιοι είπαν το χρειαζόμαστε κιόλα, ότι μα βοηθάει. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κλάδος ε, προηγείται στη φιλοδοξία σε σχέση με κυβερνήσει. το οποίο κάποιε φορέ είναι πόδινο να το βλέπει κανεί, αλλά και πάλι εφόσον καταφέραμε να πετύχουμε τη συμφωνία δεν υπάρχει πρόβλημα. τι είδου συνέχεια θα δοθεί και τι χρειαζόμαστε επεγνωσμένα. Πρώτα απ' όλα, α είμαστε ειλικρινεί. Ο στόχο δεν συνάδει με το Παρίσι είναι μια σημαντική αρχή. Υπερβαίνει κατά πολύ τα όσα συζητάει ο ΙΚΑΟ, οπότε αν τα συγκρίνουμε μπορεί ο ΙΚΑΟ να πει ότι είναι ο πρώτος ε, παγκόσμια κλάδος με συμφωνία, αλλά ο IMO λέει ναι, αλλά εμείς έχουμε συμφωνία με απόλυτη μείωση εκπομπών, με τέτοιο στόχο. Αυτή είναι η αφετηρία λοιπόν. Πρέπει να προχωρήσουμε και να αυξήσουμε το επίπεδο φιλοδοξία στους στόχους, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βελτιωθούμε σε ό,τι φορά την άμεση ανάληψη δράσης. Και εδώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, κυρία Επίτροπε, δεν ήσασταν πολύ σοφείς. Ε, συμφωνούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει το σχέδιο δράσης κτλ. Αλλά ήταν κάπως ασαφές, λίγο σαν να λέγατε εντάξει ότι αυτό θα μας απασχολεί την επόμενη πενταετία. Εμείς θεωρούμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν δράσει που πρέπει να αναλάβουμε και πρέπει να τι αναλάβουμε. Γιατί τα μόρια του διευθυντήτου, του άνθρακα βρίσκονται εκεί έξω και ε, θερμαίνουν τον πλανήτη μας. Τώρα, για το στόχο του 2030. Αν πάρουμε σοφαρά τους στόχους αυτού σήμερα, αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2030 κάθε νέο πλοίο θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, γιατί ήδη θα έχουμε τα παλιά τα οποία εκπέμπουν, οπότε τα νέα θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών. Αυτό σημαίνει ότι και η Ευρώπη θα πρέπει λίγο να σκεφτεί τι κάνει ακριβώς με όλες τις υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου, ε, γιατί αυτό δημιουργεί αυτές τις υποδομές που τελικά δεν μας, δεν μας βοηθούν να πετύχουμε το στόχο μας μέχρι το 2030. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να το εξετάσουμε στρατηγικά αυτό το ζήτημα ως Ευρώπη. Τέλος, ε, κύριε Επίτροπε, για την αεροπλοεία, τον ΙΚΑΟ, ξέρω ότι πάντα θέλετε ολοένα και περισσότερες χώρες ε, να συμμετάσχουν σε αυτή την εθελοντική φάση. Ξέρουμε όμως ότι όλη η συμφωνία ε, που ήδη ήταν αδύναμη στους στόχους της μετά την επίτευξη βλέπουμε ότι συνεχώς ε, ε, μπαίνουν παραθυράκια σε σχέση με τα προγράμματα αποζημιώσεων. Εγώ εκδηλώνω πραγματικά τον προγραμματισμό μου ε, για την αεροπλοεία και νομίζω ότι τώρα που IMO έχει πετύχει στόχους απόλυτων απόλυτη μείωση εκπομπών. Θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο και με τον ΙΚΑΟ. Ένα ε, βασικό στοιχείο θα είναι ο δικό χάρτη για το κλίμα για το 2050. Πρέπει να συμπεριλάβετε, παρακαλώ, και αυτού του δύο τομεί, ε, λοιπόν, σε αυτόν τον οδικό χάρτη για να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση και στον ΑΕΜΟ βεβαίω, αλλά ιδίω ό,τι αφορά τον ΙΚΑΟ, που θα πρέπει να τα πάει καλύτερα από εδώ και πέρα, γιατί αλλιώ είναι πολύ δυσίωνα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Προσβλέπω στη συνέχιση τη συνεργασία μας που σίγουρα θα συνεχιστεί, Ιδίω ό,τι φορά και τις εγκαταστάσεις ε, των λιμένων. Ευχαριστώ πολύ. Ποιο άλλο θα πάρει το λόγο. Ο κύριος Λίζε. Αλλά αν υπάρχει κάποιος άλλος, παρακαλώ. Κύριε Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πίτροπε. Φαίνεται να είναι αυτό ένα μεγάλο βήμα δεν το είχα ελπίσει και γι' αυτό ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, βοήθησαν στο να γίνει αυτό το βήμα. Ωστόσο, όλοι όσοι λένε ότι δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι των παρουσιών έχουν δίκιο. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε ίσως θα πρέπει να συνεχίσετε να πιέζετε προκειμένου να ενισχυθεί βήμα-βήμα η συμφωνία αυτή να αυστηροποιηθεί. Και έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όμως. Ήδη για το Μάιο είχε εξαγγελθεί η πρόταση της Επιτροπής στο EMYE, αλλά αυτό έχει αναβληθεί αλλά ε, ακόμα η Επιτροπή ε, λέει ότι δεν θέλει να υποβάλει άλλες προτάσεις από τον Ιούνιο και μετά. Θεωρούμε ότι αυτό είναι παράλογο. Εμείς επιθυμούμε να διατυπώνονται και άλλες ε, προτάσεις γιατί από τις συμβάσεις αυτές τις διεθνείς συμφωνίες απορρέουν κάποιες υποχρεώσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υποβάλλετε την πρόταση αυτή από κοινού με τους συναδέλφους αλλά και πάλι γενικά ε, στη διεύθυνση της Επιτροπής θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δυνατόν να μην ε, υποβάλλονται πλέον προτάσεις από τον Ιούνιο κλπ. Γιατί θα έχουμε μεν μια νέα επιτροπή, αλλά ευθύ εξ αρχής δεν πρόκειται να επαβάλουν προτάσεις. Άρα μπορεί να περάσουν δύο χρόνια μέχρι τις ότου να έχουμε κάποιες καινούριε προτάσεις. Δεν είναι δυνατόν όμως να έχουμε, να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια διακοπή δύο ετών, γιατί υπάρχουν κατεπήγοντα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και μετά το μήνα Ιούνιο. Ευχαριστώ. κύριε Ντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να αρχίσω ευχαριστώντα την Επίτροπο επίση. Θυμάμαι που ήμασταν εδώ, σε αυτή την εδώ αίθουσα, μαζί σα και επανέρχεστε για να μα δώσετε τι τελευταίε εξελίξει για τα όσα γίνονται στον IMO. Πρέπει να πω ότι αυτή τη φορά πρόκειται για εξαιρετικά θετικό βήμα μπροστά. Ωστόσο θα ήθελα να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Γιατί μιλάμε για το 2050, είναι μακριά. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν αλλαγές. Για μένα το 2050 είναι μακροπρόθεσμα ε, σορίζοντας. Θα πρέπει να ληφθούν όμως και βράχοι και μέσο πρόθεσμα μέτρα, ώστε ο τομέας της αυσυπλογίας να είναι στο δρόμο της μείωσης των εκπομπών ως κλάδος. Και θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσο η Κομισιόν εξετάζει μέσω και βράχει πρόθεσμα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν οι μειώσεις που θέλουμε. Ε, γιατί όταν μιλάμε για στόχους του 2050, ανησυχώ μήπω έχουμε μια μακρά περίοδο όπου τίποτα ή πολύ λίγα θα γίνουν και τελικά θα καταλήξουμε στο να λέει ο κάθε κλάδος ότι τώρα δεν έχουν χρόνο πια για να αρχίσουν να έχουν αποτελέσματα. Και να τονίσω κάτι ακόμα, ότι κάθε μεμονωμένος τομέας, κάθε μεμονωμένος κλάδος εσύ χρειάζεται να συμβάλλει γιατί αυτό, αυτά όλα ξεπερνούν την ευθύνη αποκλειστικά ενός, ενός άλλου κλάδου. Ε, δεν μπορεί οποιοδήποτε κλάδος να μην συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών, γιατί προφανώς και οι υπόλοιποι κλάδοι, που, στους οποίους αστραφούμε για συμβολή, για τέτοιες μειώσεις, θα λένε ναι, αλλά όλοι οι ε, κλάδοι πρέπει να κάνουν ε, την προσπάθειά τους. Και όντω έχουν δίκιο ότι κάθε τομέας, κάθε κλάδος πρέπει να συμβάλλει στην καθολική μείωση με εκπομπών που θέλουμε να πετύχουμε. Και γι' αυτό και χάρηκα που είπατε ότι 30 χρόνια, σε 30 χρόνια είστε πεπισμένοι πως η τεχνολογία θα εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό και εγώ πιστεύω πως η τεχνολογία αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, θα αναπτυχθεί και σε αυτό το τομέα και ε, το να έχουμε κάποιον κλάδο να αποθεί τις αλλαγές διότι πιστεύει πως αυτό μπορεί να τους κρατήσει σε μια πιο άνετη κατάσταση για την ώρα αυτό θα έχει όμως αντίκτυπο μακροπρόθεσμα γιατί δεν θα βρίσκονται στην πρωτοπορία όσον αφορά την κοινοτομία και δεν θα είναι και ανταγωνιστική κατά συνέπεια σε σύγκριση με άλλους κλάδους αλλά και σε σύγκριση με άλλες υπήρους. Θα ήθελα λοιπόν ο το τη αυσιπλοεία να συμβάλλει να είναι στην πρωτοπορία τη καινοτομία και τη τεχνολογία για τα επόμενα χρόνια. Και σίγουρα τα επόμενα χρόνια η τεχνολογία θα αναπτυχθεί, αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εμεί θα δώσουμε όθηση για βράχη και μέσω πρόθεσμα μέτρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ. Νομίζω δεν έχω άλλο να Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνση που μου δίνετε αλλά και για την πίεση που μου ασκείτε. Εγώ είμαι η πρώτη που υποστηρίζω στεναρά την άρση των αρνητικών ε, ε, ε, εξωτερικών επιπτώσεων από τις μεταφορές δεν πρέπει να δεχτούμε ως κοινωνία όλες αυτές τις ε, αρνητικές εξωτερικές ε, επιρροές ε, για να και μόνο προς χάρη κέρδους. Η χορύπανση, η ρήπανση είναι πραγματικά σοκαριστική. 24% ε, είναι η συμβολή της κυκλοφορίας μέχρι στιγμής και ε, αν δεν το μειώσουμε θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα είναι ο μεγαλύτερος ρηπαίνων η ναυσιπλοεία. Εμείς πρέπει να κάνουμε λοιπόν πολύ εντατικά τη δουλειά μας. Πρέπει διαρκώς να ενημερώνουμε για αυτές τις αρνητικούς αντικτύπους. Ε, Μόνο έτσι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να θέσουμε πιο, στο, πιο τολμηρούς στόχους. Αν δεν γνωρίζει κανείς το πρόβλημα, τότε δεν αντιδρά. Νομίζω πως η Κομισιόν ε, έχει όλο ένα και καλύτερες στατιστικές, τα μοντέλα διακυβέρνησης βελτιώνονται, προετοιμάζουμε ειδικού ορισμούς που θα έρθει σε ε, λίγες εβδομάδες, τι θα πει ακριβώς απαλλαγή από τον άνθρακα, πώς θα το μετρήσουμε και πώς θα το φέρουμε στη, στο μοντέλα διακυβέρνησης πέρα από τις στατιστικές ανάγκες ανάπτυξης και απασχόλησης. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα για να υπολογίσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο αλλά και τις εξοικονομήσεις που θα προκύψουν από τις διάφορες δράσεις για να φτάσουμε στις μηδενικές εκπομπές το 2050, ίσως και νωρίτερα. Αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει διαρκείς αναθεωρήσεις και διαρκή πίεση για τα επόμενα 30 χρόνια. Γρήγορα να ανατρέξω τα όσα με ρωτήσατε. Πρώτα, κατάλογος ε, μέτρων που θα είναι μέρη της στρατηγικής του IMO. Η δουλειά ξεκινά ήδη από τον Ιούλιο. Ε, θα δημιουργηθεί, θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας και η συνεδρίαση που προβλέπεται για τον Οκτώβριο φέτος ε, θα εστιάσει στα, σε ένα πρόγραμμα δράσης για βραχυπρόθεσμα μέτρα κάποια στοιχεία που είναι επιτάπητος και πρέπει να πω ότι δεν είμαστε πολύ δημιουργικοί και καινοτόμοι σε αυτό το κατάλογο, αλλά τουλάχιστον έχουμε κάποιες αυτές προτάσεις. Πρώτον, δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας, ε, επιχειρησιακή απόδοση των πλοίων, ε, βελτιστοποίηση ε, νομίζω θα πρέπει να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες για να βρούμε συγκεκριμένες θετικές πρόθεσμες δράσεις που να μπορέσουμε να προτείνουμε τον Οκτώβριο στην ΜΕΠΕ 73. Έχει ξεκινήσει η δουλειά λοιπόν, δεν περιμένουμε για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ε, για, την, ε, για το MRV δηλαδή εποπτεία ε, αναφορά ε, και επαλήθευση. Εδώ έχουμε προθεσμία που κάπως ε, παρατάθηκε και μόλις θα ολοκληρώσουμε το, η μελέτη αντικτύπου εδώ θα έρθουμε με προτάσεις. Είναι φάκελος του συναδέλφου Κανιέτε, αλλά συνεργαζόμαστε από αυτού για τους δύο τομείς τους δύο κλάδους και είμαι βεβαία ότι θα μπορέσουμε να, μετά το καλοκαίρι να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, sorry, I already said about the measures. Then it was a, question about Arctic, uh, Arctic and heavy fuel oil ban. Uh, MEP uh, instructed it. Για την απαγόρευση του ακατέργαστου ε, πετρελαίου στην Αρκτική θα αρχίσουμε στις αρχές του 2019, Είναι η επόμενη συνεδρίαση και με ενημερώθηκα ότι η απαγόρευση για την Ανταρκτική, για τη χρήση και μεταφορά ακατέργαστου πετρελαίου ισχύει σύμφωνα με την σύμβαση Μαρπόλ. Ήδη καλύπτεται δηλαδή η Ανταρκτική και τώρα ακολουθεί η Αρκτική. Ε, συνάδελφος Γκούτλαντ, ζητήσατε πάλι για το, ρωτήσατε πάλι για το πρόγραμμα δράσης. Θα πρέπει να σας πω ότι αναλάβαμε ε, ε, μία δέσμευση. Δεν είχαμε το χρόνο να συμφωνήσουμε για προγράμματα δράσης αυτή την εβδομάδα, αλλά είχαμε σαφή δέσμευση ότι θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε τουλάχιστον για ένα πρόγραμμα δράσης για βραχυπρόθεσμα μέτρα το φθινόπωρο. Αυτό έγινε και αυτό, ε, γι' αυτό δεσμευτήκαμε. την διάρκεια αυτής της διαπραγματευτικής εβδομάδας. Επίσης αναφέρθηκε... Ναι, έχουμε πρόκληση να αντιμετωπίσουμε τη Βραζιλία, την Αργεντινή και λοιπούς. Έχουν όμως διαφορετική άποψη. Θεωρούν πως ε, στην ουσία κάνουν, ε, διαχειρίζονται πράγματα γιατί δεν έχουν μεγάλους εφοπλιστές βλέπουν αυτή την πρόκληση από διαφορετική προοπτική και το κατάλαβα μόνο στο Λονδίνο όταν συνομιλούσα μαζί τους ε, ότι είναι τελείως διαφορετική αντίληψη ξεκινούν από διαφορετική θέση και ε, φέρνουν διαφορετικά προβλήματα στη συζήτηση. Ήδη το συζητήσαμε με τις υπηρεσίες μας για να βρούμε μια, τη σωστή προσέγγιση ε, που να έρχεται στην ε, δική τους άποψη κοντά, που είναι διαφορετική από αυτή των Ελλήνων ή άλλου εις χώρας με πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη ναυσιπλοεία. Η Σαουδική Αραβία βεβαίως και η ΙΠΑ είναι άλλη καθένας ε, ξεχωριστή περίπτωση. Αλλά η Σαουδική Αραβία πάντοτε διαμαρτύρεται γιατί να κυνηγάμε το πετρέλαιο ενώ υπάρχουν άλλες δυνατότητες για μείωση της χρήσης του άνθρακα. Και λέω ειλικρινά, δεν έχω τίποτα εναντίον του πετρελαίου. Εγώ έχω πρόβλημα με το τι βγαίνει από τα συστήματα παραγωγής, ε, πρόθεσης μάλλον, που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το πετρέλαιο που με βρίσκει αντίθετη. Ίσως λοιπόν να έχουμε και κάποιε καινοτομίε που μπορεί να βοηθήσουν, ε, να βοηθήσουν να χρησιμοποιηθεί τεχνολογία καθαρή. Και γι' αυτό και η Κομισιόν παραμένει ουδέτερη ως προς την τεχνολογία στηρίζουμε οτιδήποτε που μπορεί να οδηγήσει σε καθαρή κινητικότητα. Είμαστε ανοιχτοί για το τι θα προκύψει στα επόμενα χρόνια. Σε τρία χρόνια βλέπετε τα πράγματα αλλάζουν και για την αεροπλοεία να πω δύο λόγια που είναι ένα καλό παράδειγμα. Πριν από τρία χρόνια κανείς δεν ήθελε να ακούσει για υβριδικά αεροπλάνα, ηλεκτρικά αεροπλάνα, δεν γινόταν καμιά επένδυση και κανένα σχέδιο για κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Η Rolls Royce ήδη ανακοίνωσε πως ε, το 2030 θα έχει ετοιμάσει ένα νέο σύστημα προώθησης αεροπλάνων που θα είναι τελείως καθαρό. Όλοι οι μεγάλοι λοιπόν κατασκευαστές δουλεύουν για υβριδικά και ηλεκτρικά αεροπλάνα. Έχουμε ένα σωρό που προκύπτουν. Υπάρχει λόγος να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά ε, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως ε, παραμένουμε και ενεργούμε ως ένα οικοσύστημα, συνεχίζουμε να πιέζουμε μέσω των υψηλότερων φιλοδοξιών κάθε φορά σε ένα νέο κύκλο ε, ο IMO τώρα φαίνεται να έχει ακόμα περισσότερες φιλοδοξίες, αλλά όπως θυμάστε πριν από δύο χρόνια τον ΙΚΑΟ πέρασε εκείνη τη συμφωνία ορόσημο ε, ο ΕΜΟ είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε τέτοιες δεσμεύσεις και βλέπετε δύο χρόνια μόλις πέρασαν και είναι ακόμη πιο φιλόδοξοι. Πιστεύω ότι το μιλάμε, ότι τη συζητάμε, ε, ενημερώνουμε, ε, ε, ευαισθητοποιούμε για το πρόβλημα και μπορούν όλοι να το συζητήσουν άνετα, βοηθάει. Γι' αυτό και η επικοινωνία είναι πολύ ουσιαστική και είμαι ευγνώμων για τη θετική συνεργασία μαζί σας και πάντοτε θα είναι ευπρόσδεκτη η δική σας πίεση ώστε να βελτιωνόμαστε διαρκώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ σήμερα και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Α, κάτι ξέχασα. Παρακαλώ θυμίστε μου. Μπορεί να μην είναι σημαντικό, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι για το νέο σύστημα παρακολούθησης υποβολής εκθέσεων ε, και επαλήθευσης στο MRV ότι θα έπρεπε να υπάρξει πριν το καλοκαίρι. Ιδάλλως ε, έχουμε χάσει πολύ τον χρόνο, όπως είπε και ο κύριος ε, Λίζε. Του χρόνου έχουμε εκλογέ. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το επόμενο Κοινοβούλιο. Τα, τα δεδομένα των εμπορευμάτων όμως είναι σημαντικά. Έχουμε ολοκληρώσει την εξολόγηση δικτύπου και θα τα δώσουμε μέχρι το φθινόπωρο, είπα, φέτος. Ναι, αλλά και πάλι δεν υπάρχει χρόνος γιατί οι εκλογές είναι το Μάιο. Και όλα κάπως ε, σταματούν. Όπως και να έχει επίτροπε. Είναι θέμα διαφάνειας τα θέματα διαφάνεια μάλλον και τα δεδομένα πραγματικού φορτίου είναι θεμελιώδου σημασία στο πλαίσιο του MRV. Θα τεθεί κατά μέρο. Σε αυτή την περίπτωση έχει κερδίσει ο IMO. Και εμεί δίνουμε την εντύπωση ότι ρίχνουμε το επίπεδο φιλοδεξιών μας στο δικό του επίπεδο. Αυτό θα γίνει. Προτείνεται στην επόμενη αναθεώρηση να αφήσουμε εκτός ε, τη διαφάνεια και τα δεδομένα πραγματικού φορτίου. Όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε εντάσσονται στην αξιολόγηση τύπου. Δεν ε, μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα τι ισχύει για τα συγκεκριμένα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση δικτύπου. Αλλά θα συζητήσω αυτό το ζήτημα με τον Κανιέτα την επόμενη εβδομάδα. Δυστυχώ δεν είναι στις Βρυξέλλες αλλά θα του μιλήσω και θα δω. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να επιταχύνουμε τη διαδικασία, θα το επισημάνω λοιπόν και το ζήτημα. το ζήτημα που αναφέρατε συγκεκριμένα ε, εμπεριέχεται στην αξιολόγηση. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Να μας ξανάλθετε στο μέλλον σε ζητήματα που απασχολούν ε, όλους μας. Ευχαριστώ πολύ και για τη στήριξή σας. Τώρα θα περάσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με τους καρκίνους του πεπτικού συστήματος. Έχουμε τον Διευθυντή John Ryan από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και θα του δώσουμε πρώτα τον λόγο. Και μετά όποιος θέλει να πάρει τον λόγο, ας σηκώσει το χέρι. Παρακαλώ. Κύριε Ράγεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια σειρά διαφάνειες ε, για να βοηθήσω στην παρουσίασή μου. Χαίρομαι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνατε σε αυτήν την τελεγή απόψεων για να σας δώσω συγκεκριμένες πληροφορίες ε, για το έργο μας σε αυτόν τον τομέα. Πρώτα απ' όλα, καλό θα ήταν να έχετε μια επισκόπηση αυτής της κατηγορίας, ε, αυτού του τύπου καρκίνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τον Καρκίνο, που ε, παρέχει πληροφορίες που θα δείτε και στις διαφάνειες εδώ. Στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε ότι το 20% ε, των καρκίνων είναι καρκίνοι στο έντερο ε, τρίτος ε, πιο ε, συνήθις ε, καρκίνος είναι αυτός του παχαίου εντέρου για τους άντρες και δεύτερος πιο κοινός καρκίνος για τις γυναίκες. Δεύτερον, και πάλι είναι ο δεύτερος πιο θανατηφόρος καρκίνος αυτός του παχαίου εντέρου για τους άντρες και τρίτος για τις γυναίκες. Αν δείτε τις προβλέψεις για το 2018, βλέπουμε ότι ε, αναμένονται πάνω από 360.000 νέες περιπτώσεις ε, τέτοιου καρκίνου ε, και περίπου 150.000 θα είναι οι θάνατοι. Βλέπετε η ανάλυση των τάσεων δεν μας δείχνει ευβίωνα στοιχεία, αυξάνεται ο αριθμός των νέων περιστατικών Ταυτόχρονα, οι τάσει εθνισμότητα δείχνουν ότι τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια είναι θετικά. Παραμένει προτεραιότητα ο καρκίνο του τυχαίου εντέρου όμω ε, για την καταπολέμηση ευρύτερα του καρκίνου, γιατί βλέπουμε τη σημασία ε, του τύπου αυτού. Εδώ μπορούμε να είμαστε ελαφρώ αισιόδοξοι, γιατί βλέπουμε ότι ο καρκίνο του τυχαίου εντέρου είναι από αυτού του καρκίνου που μπορούν να προβλεφθούν. Ε, και αν υπάρχει έγκαιρη διάγνωση αυτό μπορεί να σώσει τη ζωή, να σώσει ζωές. Πέρυσι υπήρξαν ορισμένες δημοσιεύσεις που μας δείχνουν κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία και τα επισημαίνω. Βλέπετε εδώ ότι 20 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, ε, προβλέψει συγκεκριμένα σε σχέση με το 2012 που δημοσίευθηκε πρώτη ε, έκθεση. Από τις 10 χώρες λοιπόν πέρασαμε στις 20 που κάνουν δηλαδή έλεγχο στον πληθυσμό τους. Περίπου 150 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες ε, από τα 50 74 έτη τους, τα κρατημέλη, στοχεύονται μάλλον από αυτό τον διαγνωστικό έλεγχο. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Δείχνει ότι υπάρχει ανωδική τάση στον αριθμό των ανθρώπων που καλύπτονται από τον έλεγχο. Όμω, η υλοποίηση αυτών των ελεγκτικών προγραμμάτων ενδιαφέρει από χώρα σε χώρα. Ε, συμπεριλαμβανομένου και το πρωτοκόλλο που ε, ακολουθείτε για τις εξετάσεις. Απαιτούνται λοιπόν, ε, απαιτείται συνέχιση των προσπαθειών σε αυτό το τομέα. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τις εφημερίδες τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά είχαμε τεράστια σκάνδαλα σε δύο κρατημέλη σε σχέση με τον ποιοτικό έλεγχο στα ε, προγράμματα καρκινικού ελέγχου. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που δείχνουν ότι απαιτούνται βελτιώσεις ε, και ορισμένα κενά θα πρέπει να καλυφθούν. Εφόσον αναμένεται σημαντική αύξηση των περιστατικών ε, του καρκίνου, του παχαίου συντέρου και του ορθού εξαιτία τη γύρανση του πληθυσμού, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων ε, διαγνωστικού ελέγχου. Εμείς προτείνουμε τρεις ε, πρωτοβουλίες. Πρώτον, έχουμε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του καρκίνου με έναν κατάλογο 12 τρόπων ε, περιορισμού του κινδύνου να πάθει κάποιος το καρκίνο αλλά και πιο συγκεκριμένα τον για να αποφύγει τους καρκίνους ε, του εντερικού συστήματος και με, αποφύγει του καπνίσματος, του αλκοόλ και τα γνωστά. Ε, αλλά έχουμε και την, ε, τον εμβολιασμό των παιδιών κατά της υπατήτητας Β, αλλά και την οργανωμένη συμμετοχή σε προγράμματα διαγνωστικού ελέγχου. Θα χρηματοδοτηθούν και από μια νέα κοινή δράση υπό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Υγείας που ξεκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο αφορά την ε, τεχνική αρρωγή. Ε, για δύο χώρες ε, το έχουμε διοργανώσει. Αυτή η τεχνική αρρωγή χρηματοδοτείται από τον ενωσιακό προπολογισμό. Αυτή τη στιγμή εντοπίζουμε τις χώρες που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια και μετά την οργανώνουμε. Και υπάρχει μια άλλη πρωτοβουλία για την βελτίωση της ποιότητας της διάγνωσης και της περίθαλψης. Αναπτύσσονται ε, συστάσεις και κατευθυντήρες γραμμές που θα είναι διαθέσιμες για ασθενείς ε, και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και για τους επαγγελματίε της υγείας. Σε ό,τι αφορά ε, τις μη μεταδοτικές ασθένειες αλλά και τις τους καρκίνους ε, του γαστροεντερικού συστήματος. Βλέπουμε ότι έχουμε και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που μας δίνουν στόχο βελτίωσης και αυτό είναι κάτι το οποίο, στο οποίο, το οποίο έχουν προσυπογράψει και τα κράτη-μέλη από κοινού με την Επιτροπή. Οπότε θέτουμε αυτούς τους διεθνείς ε, στόχους ως ε, σημείο αναφοράς σκοπεύουμε να εντοπίσουμε και να υλοποιήσουμε βέλτιστες πρακτικές ή επεμβάσεις ή ε, παρεμβάσεις που έχουν αποδειχθεί επιτυχία στο παρελθόν. Και θέλουμε να αυξήσουμε τον κατάλογο αυτών των ε, βέλτιστων πρακτικών και παρεμβάσεων που βλέπουμε ότι έχουν θετικό αντίκτυπο η Επιτροπή θέλει να στηρίξει την υλοποίηση αυτών των ε, πρωτοβουλίων σε εθνικό επίπεδο και μέσω του ανοσιακού προπολογισμού και μέσω άλλων ε, χρηματοδοτικών μηχανισμών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε κρατημέλη σε εθελοντική βάση έχουν επιλέξει τον τομέα των διαγνωστικών ελέγχων του καρκίνου του παχαίου εντέρου και του ορθού για να κινητοποιήσουν προγράμματα σε εθνικό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τα κράτη-μέλη για να εντοπίσουν τους τομείς στου οποίους θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο. Και ξεφεύγουμε από τα όρια των συνήθων εταίρων, γιατί πρόσφατα, για παράδειγμα, η Εταιρική Τράπεζα Επενδύσεων μας ζήτησε να τη βοηθήσουμε για την επιλογή κριτηρίων συγκεκριμένων θεραπευτικών κέντρων για να επενδύσει η τράπεζα σε τέτοια θεραπευτικά κέντρα. Οπότε αποκινούμε τα κράτη-μέλη εξετάζουμε τους εθνικούς στόχους και προσπαθούμε να επιλέξουμε συγκεκριμένα προγράμματα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, δυσμενείς συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ε, τα συστήματα υγείας, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το γνωρίζετε σαφώ, ότι υπάρχει ζήτημα γύρανση του πληθυσμού, χρόνιε παθήσει, αυξανόμενη ζήτηση για την υγειονομική περίθαλψη, νέε και δαπανηρέ ε, θεραπείες και τεχνολογίε ε, και όλα αυτά με περιορισμένους ε, υγειονομικούς πόρους. Γι' αυτό απαιτείται μεταρρύθμιση των υγειονομικών συστημάτων για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση της υγείας και στην πρόληψη και εδώ μπαίνει και το θέμα του διαγνωστικού ελέγχου Ελπίζουμε επίσης ότι η ανάλυση που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον ΟΣΑ και το Παρατηρητήριο Υγείας, καθώς και οι εθνικές εκθέσεις, τα εθνικά προφίλ, θα μας εντοπίσουν τυχόν κενά και θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το εθνικό σχέδιο καρκίνου. Έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή και Φυσικά συνεχίζουμε την προσπάθεια και με τα Μητρώα, γιατί αυτή είναι σημαντική πτυχή. Να έχουμε δηλαδή ευρωπαϊκά, ποιοτικά ευρωπαϊκά Μητρώα, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Διευθυντά, συνάδελφοι, ε, μπορείτε να βάλετε ερωτήσεις. και Σπότσου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε γιατί έχω πλήρη επίγνωση της προσήλωσής σας σε αυτό το τομέα. Εκτιμώ πολύ το έργο της Επιτροπής όσον αφορά τον καρκίνο του εντέρου και του ορθού. Και σήμερα μιλούμε για καρκίνους του εντερικού συστήματος και οι παρατηρήσεις μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί προκαλούν 365.000 περιπτώσεις θανάτου στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι χίλια άνθρωποι ε, αποθνίσκουν ε, ημερήσίως από αυτό τον τύπο καρκίνου αν σκεφτούμε ποιος είναι ο αριθμός των θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων ή αεροπορικών ε, δυστυχημάτων, βλέπουμε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός. Ε, δεύτερον, έχουμε έναν εχθρό σε αυτό το πεδίο, ο, το καρκίνο του Παγκρέατος πολλές μορφές καρκίνου μπορούν να προληφθούν, όπως ο καρκίνος του εντέρου, με διαγνωστικούς ελέγχους ή μπορούν να θεραπευθούν. Αυτό δεν γίνεται με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες για τη διάγνωση αλλά και για τη θεραπεία. Αυτή τη στιγμή διαγνωστεί πάντα είναι υπερβολικά αργά. Άρα ο καρκίνος στο πάνγκρεας ε, ισοδυναμεί μια θανατική καταδίκη. Τώρα, 64% των Ευρωπαίων ε, λένε ότι δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Είναι η πιο θανάσιμη μορφή καρκίνου, θανατηφόρα, με 3% ε, ε, ποσοστά επιβίωσης και για 5 χρόνια ενώ ο καρκίνος του πνεύμονα είναι 12%. Τα ποστά επιβίωση για τις περισσότερες μορφές ε, καρκίνου έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι για το καρκίνο στο πάγκρεας. Το 2025 ε, θα έχουν αυξηθεί τα κρούσματα καρκίνου ε, και η διάγνωση είναι πολύ δύσκολο να γίνει στα πρώιμα στάδια. Ο βασικός λόγος ακριβώς για την ε, μη ε, θεραπεία είναι η αδυναμία έγκαιρης ε, διάγνωσης. Και είναι άρα λοιπόν ζωτική σημασία οι, περισσότε... οι ασθενείς να έχουν μια έγκαιρη διάγνωση. Ε, Βεβαίω γνωρίζουμε ποια είναι τα στοχευμένα μέτρα που απαιτούνται για μια πρώιμη διάγνωση και θεραπεία καρκίνου στο πάγκρεας, αύξηση της ε, ερευνητική δραστηριότητας στο επίπεδο της πρόληψης και εργαλεία πρώιμης ανείχνευσης και νέες ε, αποτελεσματικές θεραπείες. Αναφερθήκατε στην συγκέντρωση των δεδομένων. Σας ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας. Ε, χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε σχέση με την έγκαιρη διάγνωση, τα συμπτώματα και ε, αυτές τις μορφές καρκίνου και βεβαίως ε, αποτελεσματικές αντιδράσεις από τις χώρες μέλη. Το ερώτημά μου είναι πώς προτίθεστε να πετύχετε τους στόχους σας για τον καρκίνο γενικά και ιδιαίτερως για τον καρκίνο στο πάγκρος, Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιώργο ε, Είμαι ενθουσιασμένη που μπορούμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που πραγματικά βρίσκεται, ε, απασχολεί τόσο πολύ τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Ο καρκίνος, η καρκίνοι του εντερικού συστήματος μας απασχολούν, δίνεται έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση κλπ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτή τη μορφή καρκίνου. Αλλά θα πρέπει να καταφέρουμε να αποδραματοποιήσουμε όλα αυτά, γιατί πολλοί από τους συμπολίτε μας στην Ευρώπη ε, φοβούνται σχεδόν τη διάγνωση. Άρα λοιπόν είναι απρόθυμοι να κάνουν κάποια προληπτική εξέταση. Άρα λοιπόν, πώς ε, θα μπορούσαμε να αποδραματοποιήσουμε όλη την κατάσταση ώστε να παροτρύνουμε τον πληθυσμό να προβεί σε διαγνωστικούς ελέγχους. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτω. Από την άλλη, μας είπατε, εάν κατάλαβα καλά, πέντε χώρες μέλη ζήτησαν μία βοήθεια από την ε, κοινότητα μέσω του προγράμματος για την υγεία. Όταν βλέπουμε όλη την εργασία που πρέπει να γίνει για τους καρκίνους ε, θα πρέπει να δούμε, έχουμε επαρκή σπόρους. Αυτή τη στιγμή συζητούμε όλοι για το μελλοντικό δημοσιονομικό πρόγραμμα και ε, κάθε φορά η υγεία είναι ο φτωχός ε, συγγενής. Σήμερα το πρωί είδα ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία τοποθεί την υγεία στο επίπεδο της ένταξης των μεταναστών. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως σοκαριστικό. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Γνωρίζω ότι γίνονται κάποια διαβήματα στο πλαίσιο της Επιτροπής μας, αλλά θα πρέπει πράγματι να καταφέρουμε να ασκήσουμε καλύτερη πίεση στον προπολογισμό προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συμπολιτών για αυτό το πρόβλημα του καρκίνου, όχι μόνο του καρκίνου του εντέρου, αλλά του καρκίνου στο πάγκρας για παράδειγμα. Υπάρχουν και οι όγκοι στον εγκέφαλο, υπάρχουν οι παιδιατρικοί καρκίνοι, οι καρκίνοι στα παιδιά. Άρα υπάρχει τόση δουλειά να γίνει και οι απαντήσεις που θα μπορούσαν να θα έδειχναν την προσθέμενη αξία στα μάτια των Ευρωπαίων συμπολιτών μας. Άρα λοιπόν, θεωρείτε ότι είναι επαρκή η χρηματοδότηση που προβλέπετε για την υγεία. Εγώ πιστεύω πως όχι. Και πώς θα μπορούσαμε να παροτρύνουμε περισσότερο τους συμπολίτε μας να συμμετάσχουν στους ε, προληπτικούς ε, πρώιμους διαγνωστικούς ελέγχους χωρίς να έχουν αυτό το δρόμο να διαγνωστούν που τους κάνει πρόθυμους. Η κυρία Ντάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή που βρίσκεται εδώ και χαίρομαι που συζητούμε το θέμα αυτό γιατί είναι η δεύτερη πιο συνήθιση αιτία θανάτου μετά από τον καρκίνο του πνεύμονα και του στήθους γιατί ε, σε σχέση με τους, ε, βιώσ... με τους στόχους της βιώσιμης ε, ανάπτυξης που έχουν προσυπογράψει οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η... η καταπολέμηση του καρκίνου δεν καλύπτει την, πράληψη, την πρόληψη. 8% δαπανώνται για την θεραπεία, αλλά μόνο 3% για την πρόληψη του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε αυτά τα νούμερα, γιατί εμείς ε, ως ε, πολιτικοί φορείς θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει εδώ κάποια πρόοδος. Γιατί οι περισσότεροι καρκίνοι είναι προβλέψιμοι εάν προσθέσουμε εδώ το, την ποιότητα διαβίωσης, ε, τα ποσοστά κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα κλπ. Και ε, βεβαίως ε, ένας υγιής τρόπος διαβίωσης δεν επαρκεί. Θα πρέπει να θεσπιστεί από εμά μια έγκαιρη πολιτική πρόληψης μέσω πρώιμων διαγνωστικών ελέγχων. Οι καρκίνοι του εγκαίρου δεν εξαρτώνται από την ηλικία υπάρχουν κάθε χρόνο 6.000 ε, νέα περιστατικά και αυτή τη στιγμή ε, τα συστήματα ε, διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται σε, γίνονται σε εθελοντικό επίπεδο. Υπάρχουν χώρες μέλη που σε άλλες χώρες έλεγχοι που γίνονται στα 30, άλλες στα 60, άλλες στα 50 κλπ. Ε, που σε ορισμένε περιπτώσει είναι ίσως υπερβολικά αργά. Η εξέταση έπρεπε, ε, σύμφωνα με τους ειδικού να ξεκινήσει από τα 45 έως τα 49. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ευέλθιστες πρακτικές, ούτως ώστε ε, στο μέτρο του δυνατού οι χώρες μέλη να μπορέσουν να εναρμονίσουν την επιλεξιμότητα για τα προγράμματα διαγνωστικού ελέγχου και να ξεκινούν σε μία ηλικία όπου η ανείχνευση μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική θεραπεία. Σας ευχαριστώ. Εάν όχι. Well, thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ερωτήσεις Επιτρέψατε μου να σας πω ότι έχει γίνει σε ερευνητικό επίπεδο όσον αφορά το καρκίνο του εντέρου. Έχω κάποια στοιχεία, παρόλο που δεν λένε πολλά αυτά καθ' αυτά. Στο πλαίσιο του προγράμματος 7, 15% του συνολικού αριθμού ε, αφιερώθηκαν στον καρκίνο του εντέρου. 1,5 δισεκατομμύρια του προγράμματος δαπανήθηκαν για τον ε, καρκίνο του εντέρου. Ε, και, συγγνώμη, 15% από αυτά στον καρκίνο του εντέρου. Και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ε, στην ανάπτυξη του καρκίνου ως ε, ε, αποτέλεσμα was, του από το βακτηρίδιο κόλλη. Ε, 14% των χρημάτων για τον καρκίνο δίνονται και πάλι εδώ για, για τον καρκίνο του εντέρου Όσον αφορά τους μηχανισμούς διαγνωστικού ελέγχου, ε, υπάρχουν smartphone τα οποία ελέγχουν την αναπνοή των ε, ασθενών ή υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης κάποιων μικροβίων στον, ε, στο στομάχι για να έχουμε κάποιες βιοδείκτες για την ανείχνευση του καρκίνου, του εντέρου. Συνήθως το πρόβλημα, ωστόσο, δεν, ε, τοποθετείται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, αλλά στο επίπεδο των χωρών μελών. Και απαντώντα στα όσα είπε η κυρία Γκροστέτ σε σχέση με το κατά πόσο τα χρήματα είναι αρκετά, θα έλεγα ότι είναι μια ερώτηση δύσκολο να απαντηθεί γιατί έχω συγκεκριμένα παραδείγματα όπου δόθηκαν χρήματα στις χώρες μέλη και στη συνέχεια οι χώρες δεν μπορούσαν να τα ε, δαπανίσουν. Άρα τα ποσοστά παρόφησης των χωρών που βρίσκονται στη μεγαλύτερη ανάγκη προκειμένου να βελτιώσουν τα ε, προγράμματα εξετάσεων τα ποστά απορρόφησης από τα ιατρικά Ινστιτούτα, τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία είναι περιορισμένος. Γι' αυτό είχαμε την ιδέα να τους ε, δώσουμε στη διάθεσή τους εμπειρογνώμονες προκειμένου να τα σχεδιάσουν καλύτερα αυτά τα προγράμματα εξετάσεων και να τα βελτιώσουν. Ε, προσπαθήσαμε να αναγνωρίσουμε τις χώρες που χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να μεταβούν εκεί οι εμπειρογνώμονες. Δεν προσπαθούμε να θεσπίσουμε ε, νέες στρατηγικές, αλλά προσπαθούμε να συνεργαστούμε τις χώρες μέλη για να αναγνωρίσουμε, να ανοιχνεύσουμε τις ανάγκες προκειμένου να ενεργοποιηθούν και οι αντίστοιχοι πόροι του προπολογισμού για να τις στηρίξουμε. Για μένα λοιπόν δεν είναι κατά πόσο επαναληπτή πόρη στο πρόγραμμα έρευνα κλπ. Αλλά το πρόγραμμα είναι πώ μπορούμε να μεταφράσουμε τα χρήματα αυτά σε κάτι πραγματικά ένα αποτελεσματικό επιτόπου. Ε, γι' αυτό προσπαθήσαμε πραγματικά να, στη συνεργασία με τι χώρε μέλη να αναγνωρίσουμε τι ανάγκε προτεραιότητα και στη συνέχεια να αναπτύξουμε προγράμματα βοήθεια προσαρμοσμένα στην κάθε χώρα όχι και τα 28 μέλη, αλλά πέντε ή έξι που χρειάζονται καταπηγόντως βοήθεια. Όταν η εξι που χρειαζονται καταπηγώντας Γκροστέτ ε, αναφέρθηκε στο ζήτημα της αποδραματοποίησης των εξετάσεων προκειμένου να μην υπάρξει αρνητικό αποτέλεσμα, αυτή είναι μια δύσκολη συζήτηση γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει επαρκής ε, εκπαίδευση, διαφώτιση του πληθυσμού και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Χρειάζεται ε, ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βελτιώσει τη συνειδητοποίηση της ανάγκης υποβολής εξετάσεις. Για παράδειγμα για τον ιό του AIDS ήταν πολύ δύσκολο για τους πολίτες να πάνε να κάνουν αυτές τις εξετάσεις γιατί γνώρισαν τους οδυναμοί με μια θανατική καταδίκη. Αλλά αυτή τη στιγμή ε, τώρα πια ε, είναι μια ε, σηματοδοτεί την θεραπείας όχι τη θανατική καταδίκη το AIDS. Άρα λοιπόν θα πρέπει και το ιατρικό σώμα να κάνει κάποια πράγματα. Γι' αυτό ε, δαπανούν πολλά χρήματα για τον κώδικα του καρκίνου προκειμένου να μειωθεί το αλκοόλ, να σταματήσει το κάπνισμα και να γίνονται εγκαίρως εξετάσεις. Και εάν οι χώρες μέλη μπορούν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στους ε, πολίτες, τότε σαφώς θα βελτιωθούν οι στρατηγικές πρόληψεις. Τώρα, σχέση με τα όσα είπε η κυρία Νταλή για τους ε, διάφορους ε, τύπους εξετάσεων, θα ήθελα να πω το εξή. Έχουμε μια βασική γραμμή όσον αφορά τη στάσης για τον καρκίνο που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών για τρει τύπου. Ε, του εγκεφάλου, του στήθους ε, και του εντέρου και ορθού. Και εκπονήσαμε τρεις εκθέσεις σχέση με το πώς μπορούν να εφαρμοστούν στις χώρες μέλη. Και ε, περάσαμε από 10 στις 20 χώρες. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στην ηλικία και στις μεθόδους ανείχνευσης καθώς και ε, τον έλεγχο ποιότητας. Γι' αυτό επενδύσαμε και σε ένα κοινό ερευνητικό κέντρο για να βελτιωθεί ο έλεγχος ποιότητας σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα, γιατί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού, ε, για παράδειγμα σε δύο χώρες μέλη που τελικά κατέληξαν σε σφαλμένες, καταλήγουν σε σφαλμένες διαγνώσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στις χώρες μέλη, να επηρεάσουμε την κατάσταση μέσω των εμπειρογνωμόνων που προσπαθούν να διαμορφώσουν πιο αποτελεσματικά τους διαγνωστικούς ελέγχους δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας ότι το... οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών των ασθενών είναι τεράστιες. Και στο επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα, γιατί συνεχίζει να παραμένει μια προτεραιότητα, ενασχόληση με αυτές τις νόσους ε, Συμφωνώ ότι οι τύποι αυτοί καρκίνου τελικά, οι αρρώστιες αυτές, οι νόσοι αυτές είναι παραμελημένες ε, νόσοι που έχουν κάπως παραμεληθεί από την ε, χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Τελευταίο σημείο τώρα στην ημερήσια μας διάταξη για σήμερα είναι κοινή συζήτηση για το τροπο, γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς 1507-810 και γενετικός τροποποιημένος αραβόσιτος που συνδυάζει δύο ή τρεις από τις μεμονωμένες σειρές που προανέφερα και ο τροποποιημένος αραβόσιτος GA21. Uh, usually we start with the co-sponsors. Uh, Να δούμε ποιος είναι εδώ. Η κυρία Μπόιλαν, παρακαλώ πείτε μας τα. Σας ευχαριστώ. Οι συνεισηγητές δεν είναι εδώ γιατί παλιότερα έχουμε ξανασυζητήσει επανελειμμένα το θέμα ε, τόσες πολλές φορές. Η διαδικασία της ένστασης είναι μακρά και συνεχιζόμενη. Ε, η ένστασή μας βασίζεται στην ίδια, στα ίδια επιχειρήματα. Ε, είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα. Έχουμε ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες. Λέμε ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Το ψήφισμα αυτό και τα προηγούμενα δηλώνουν σαφώς ποια είναι η αντίρρησή μας. Οι γενετικω τροποποιημένοι οργανισμοί είναι αντίθετοι με την κινητική νομοθεσία και πρέπει να αλλάξουμε μέχρι ότου να έχει αναθεωρηθεί αυτή, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά τα προβλήματα δημοκρατικής νομιμότητας της απόφαση ε, που η ίδια η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει. Καλούμε λοιπόν την ε, Επιτροπή να στηρίξει τις δεσμεύσεις για την βιολογική ποικιλομορφία και να, ε, ε, να σταματήσει τη χρήση των σειρών που είναι ανθεκτικές στην γλυφοσάτη. Έχουμε μια τακτική έκθεση στα ζανιοκτώνα αυτά ε, και ε, που, τα οποία οδηγούν και σε σοβαρή υποβάθμιση του εδάφους. Ε, έτσι υπονομεύουν το μελλοντικό δυναμικό του εδάφους. Ωστόσο, η έστασή μας ε, στηρίζεται και στο, στο ότι κανονικά μπορούμε να δούμε όλα τα διαθέσιμα ε, παρατήματα σε σχέση με τη διαδικασία περί γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, αλλά αυτά δεν υπάρχουν ε, στο, στο site του ΕΦΣΙ και άρα δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε και τις αναφορές από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Άρα λοιπόν δεν έχει καλωθηθεί η διαδικασία όπως έπρεπε. Αυτά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Από τους υπόλοιπους συνεισηγητές δεν βλέπω κανέναν άλλον. Ποιο θα ήθελε το λόγο για αυτό το θέμα, για αυτές τις ενστάσεις, τις αντιρρήσεις. Ίσως η κυρία Γκέρλινγκ. Μάλιστα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ τον συνάδελφο κύριο Φιώνα ονόματος του ΕΛΚ. Θα ήθελα να πω ότι το ΕΛΚ διαφωνεί ε, με την πρόταση ψηφίσματος. Και θα πούμε βέβαια τα ίδια που λέμε πάντα, αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι. Η ΕΦΣΑ έχει εξολογήσει στο παρελθόν αυτό τον αραβόσιτο και είχε εκφράσει θετική γνώμη το 2017, δεν είχε εντοπίσει ε, ανησυχίες για την υγεία και κατέληξαν ότι ήταν εξίσου σε αυτοί οι οργανισμοί σε σχέση με τους συμβατικούς ε, ε τύπους. Επίσης δεν υπάρχει ε, νομική βάση αυτή. Ε, υπάρχουν πολλές αναλυθείς, πολλοί αναλυθείς ισχυρισμοί. Στην παράγραφο ε λέει ότι αποδεικνύεται ότι ε, οδηγούν σε υψηλή χρήση βλαβερών ζυζανιοκτώνων, όμως δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτόν τον ισχυρισμό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια παραπομπή όταν έχουμε τέτοιου ισχυρισμού. Βάσει αυτού του ισχυρισμού καταλήγεται στην παράγραφο F ότι οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί ε, θα εκτίθενται στη γλυφοσυνάτη σε υψηλότερη συγκέντρωση. Και πάλι λοιπόν γίνονται ισχυρισμοί ε, χωρίς να τεκμηριώνονται. Συμφωνήσαμε επ' ενός κανονισμού για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, βλέπουμε ότι ε, τηρεί τους κανόνες δεν υπάρχει κάτι που να αποδεικνύει το αντίθετο και η ΕΦΣΑ καταλήγει ότι το, ο μεταραγμένο οργανισμό είναι ασφαλή. Πρέπει λοιπόν να εμπιστευτούμε την υποστημονική τη γνώμη. Ιδάλω, αν δεν το κάνουμε για πολιτικούς λόγους, τότε αυτό είναι πρόβλημα γιατί γίνεται μια πολιτική διελκυστίνδα. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ακολουθούμε τα επιστημονικά δεδομένα που αυτό είναι δυνατόν και σίγουρα σε αυτή την περίπτωση είναι. Υπάρχουν πολλά στοιχεία Όλα έχουν ληφθεί υπόψη από την ΕΦΣΑ, στην οποία δαπανούμε πολλά χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ακριβώς για να κάνει τέτοιου είδους επιστημονικές ε, αξιολογήσεις και δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να την διαψεύσουμε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Φιέλνερ καλεί τα μέλη να καταψηφίσουν την πρόταση. τα ίδια ζητήματα ισχύουν, δεν χρειάζεται να τα να επεκταθώ περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο. Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως να ακούσουμε τα ίδια επιχειρήματα για από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα είμαστε να τον πιο σύντομοι. Έχουμε να κάνουμε εδώ δύο ψηφίσματα, ένα για νέα διοδότηση και ένα για ανανέωση και για τα δύο η ΕΨΑ έχει κάνει σε βάθος αξιολόγηση κινδύνου για τη νέα διοδότηση και για την ανανέωση και οι δύο καταλήγουν ε, σε θετική γνώμη, όπως ανέφερε και ένα μέλος του Κοινοβουλίου. Τα κράτη-μέλη έχουν όντως ε, σχολιάσει τις αιτήσει και η ΕΦΣΑ έχει ε, εξηγήσει τη θέση τη στα σχόλια και κατά τη διάρκεια μια συνεδρίασης και ε, το ευρύ κοινό έχει δυνατότητα να υποβάλει σχόλια στι νομοδοτήσει τη ΕΦΣΑ και η ΕΦΣΑ κατέληξε ότι από τα δημόσια σχόλια δεν προέκυψαν νέε επιστημονικέ πληροφορίε, επιβεβαίνονται λοιπόν η θετική γνώμη και διευκρίνησε ότι τα, κρατη τα σχόλια που έλαβε από τα κράτη-μέλη δεν έχουν τροποποιήσει τη θετική γνώμη. Βάσει τούτου, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη να διοδοτήσουν ε, ε, την, ε, την πρώτη αίτηση και να ανανεώσουν τη δεύτερη. Αυτό έγινε στις 21 Απριλίου, τότε το συζητήσαμε δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια γνώμη ούτε υπέρ ούτε κατά. Γι' αυτό και υποβάλαμε ε, χθες στην Επιτροπή Ενστάσεων και πάλι δεν υπήρχε κάποια γνώμη. Εν συντομία λοιπόν η Επιτροπή δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να απορρίψει ε, αυτές ε, τις αιτήσει γιατί έχουμε ακολουθήσει πλήρως και κατά γράμμα τη διαδικασία. Δεν έχουμε ξεφύγει καθόλου από τα όσα προβλέπονται στους κανόνες. Πράγματι, το δικαίωμα κοινοβουλευτικού ελέγχου ε, έγκυται στο κατά πόσο η Επιτροπή υπερβαίνει τις εξουσίες της ή όχι και επί της αρχής ούτε καν απαιτείται να σχολιάσουμε τα υπόλοιπα που αναφέρει το Κοινοβούλιο. Φυσικά, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε τυχόν παρατηρήσεις, όπως η έκκληση αναστολής του σχεδίου απόφασης, έκκληση για νέα απόφαση που έχει απορρίψει ε, το Κοινοβούλιο και ζήτησε από την Επιτροπή να κάνει νέα πρόταση. και αν υιοθετηθεί κάτι καινούριο μπορούμε να το σχολιάσουμε. Ευχαριστώ. Ωραία, φτάνουμε στο τέλος Τη σημερινή συνεδρίαση. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες της 9. Γεια σας.